Λοιπόν, θα ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί αργούμε, αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Ε, όμως ε, πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε διότι θα κάνουμε πρώτη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, του Σέρτζο ε, Κοφεράτη σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική απασχόληση. Πρόκειται για μια έκθεση ε, για την οποία επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε και που επαναλήφθηκε και συζητήθηκε και σήμερα το πρωί, είναι η κοινή οργάνωση κάποιων πολιτικών που σχετίζονται με την μετανάστευση. Στόχος μας εδώ και της Κομισιόν βεβαίως είναι να υπάρξουν διατάξεις σωστές έτσι ώστε ένα από τα πιο ασθενή τμήματα της αγοράς, δηλαδή οι εποχικά απασχολούμενοι, να ε, έχουν σαφώς ορισμένες προϋποθέσεις, τρόπους εφαρμογής ε, και δικαιώματα ορθώς αναγνωριζόμενα. Έτσι ώστε στην ουσία αυτός ο εποχικός ε, απασχολούμενος να είναι ισότιμος με τους άλλους ε, εργαζόμενους. Μαζί με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ευχαριστώ βεβαίως κυρίως τον συνάδελφο Μωράης αλλά και ολόκληρη την Επιτροπή που ε, άκουσε προσεκτικά τις παρατηρήσεις μου σήμερα το πρωί. Ξεκινήσαμε λοιπόν μαζί με τη ΛΥΜΠΕ αυτήν την ε, εργασία, ε, συνεργαζόμενοι στενά, γιατί θεωρώ ότι και τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά και η μεθοδολογία συνεργασίας θα πρέπει να είναι σαφής και για το μέλλον. Στην ουσία έχουμε να πούμε τα εξής. Πρώτον όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής. Για πάρα πολύ καιρό η εποχική απασχόληση είχε ε, περιγραφεί με τρόπο εξαιρετικά ελαστικό. Με στόχο τελικά να ε, αφαιρεθεί από τους εργαζόμενους ένα μεγάλο κομμάτι της προστασίας το οποίο δικαιούντο. Για τον λόγο αυτό η εποχική απασχόληση πολύ συχνά, από υπερβολικά συχνά μάλλον, αποτέλεσε αντικείμενο κοινωνικού ντάμπινγκ, καθώς επίσης ε, και στρεβλωμένου ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καθορίσουμε τι εννοούμε εποχική απασχόληση. Δεύτερον, να δούμε το πεδίο εφαρμογής. Θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο να δώσουμε μία γενική περιγραφή ε, του τι είναι η εποχική απασχόληση και όμως μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά ε, του πεδίου εφαρμογής. Λέγοντας ότι οι διατάξεις θα πρέπει να αφορούν τη γεωργική εργασία, ε, τα ε, μποστάνια, λαχανοκαλλιέργειες, προκυπευτικά και τον τουρισμό. Και βεβαίως θα πρέπει φυσικά ε, να ε, υπάρξουν και ε, συγκεκριμένες διατάξεις εθνικές, όμως που θα βασιστούν σε μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων της κάθε χώρας. Έξι μήνες προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτούς τους μήνες και μάλλον σε αυτήν την ε, περίοδο ε, αναφέρονται και οι αρχές ε, τις οποίες ανέφερα και προηγουμένως, δηλαδή τις κοινωνικές αρχές. Η ίδια αμοιβή για ίδιες συνθήκες εργασίας. Συνθήκες εργασίας που περιλαμβάνει βεβαίως το ωράριο, το είδος εργασίας και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις συλλογικές συμβάσεις. Δεν θελήσαμε σκόπιμο να αναφέρουμε συγκεκριμένα και αναλυτικά τι σημαίνει και τι πρέπει να περιλαμβάνει η συλλογική διαπραγμάτευση, γιατί αυτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Απ' την άλλη πλευρά και για να έχουμε αξιοπρεπείς, ε, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για ανθρώπους που ζουν ε, στις χώρες μας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά επιστρέφουν στην χώρα τους, γιατί λέω εδώ εν παρόδο ότι ε, ο σκοπός είναι να φύγουν μετά οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν ε, στην χώρα τους, δηλαδή να μην έρθουν εδώ για μια συγκεκριμένη απασχόληση και μετά να παραμείνουν εδώ. Θέλουμε λοιπόν να αποθαρρύνουμε οποιαδήποτε μορφή κρυφής, λαθρέας, μαύρης ας πούμε εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι τα άτομα αυτά, οι απασχολούμενοι αυτοί, θα πρέπει να, τους δω, να, να έχουν τις δυνατότητες κινητικότητας, αλλά κυρίως θα πρέπει να τους δώσουμε ε, και ένα αξιοπρεπές κατάλημα. Ε, υπάρχει ο ορισμός του αξιοπρεπούς καταλήματος ε, των Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, οι ίδιες ε, συνθήκες ε, εργασίας και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, θεωρώ ότι είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα έτσι ώστε να υπάρχει έτσι η ισοδίκαιη μεταχείριση των απασχολούμενων, των γηγενών και αυτών των ξένων ε, εποχικών απασχολούμενων. Ο στόχος ενδεχομένως είναι φιλόδοξος, αλλά κατά την άποψή μου ε, είναι σίγουρα δεσμευτικός, αλλά ε, ε, βεβαίως θα δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως μπορούμε να προβλέψουμε και μία ενδιάμεση διαδικασία έτσι ώστε να νομιμοποιηθούν αυτοί που βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και που αυτή τη στιγμή ακόμα δουλεύουν σε μαύρη εργασία, είτε εποχική είτε όχι. Δηλαδή, η οδηγία για την εποχική απασχόληση θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά ε, να ε, ξεπεράσουν την παρανομία και να μπουν σε μια νόμιμη διαδικασία. Αυτό το ε, είπαμε και με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Κάτι άλλο. Τώρα, η ενίσχυση ε, η ενίσχυση της νομιμότητας ε, και η αποτροπή της παρανομίας ε, που, και της μαύρης εργασίας που προκαλεί, όπως είπα και προηγουμένως, συνθήκες κοινωνικού dumping, είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει. Δηλαδή, εάν υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες, τότε ο επιχειρηματίας δεν θα παίρνει πλέον, δεν θα προσλαμβάνει πλέον ε, εργαζόμενους ε, παράνομους. Θα πρέπει επομένως να μπορούμε να παρακολουθούμε και να κάνουμε ελέγχους από τους ελέγχους που θα κάνει το κράτος για την είσοδο των ατόμων αυτών ε, ε, μέχρι ε, το, τις συνθήκες εργασίας, τις συνθήκες που εγώ ονομάζω συνθήκες του, του, πολίτη, δηλαδή σωστό κατάλημα, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και γενικότερα εφαρμογή οτιδήποτε περιέχεται στις συλλογικές συμβάσεις. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος λοιπόν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και της εργασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ότι η εποχική απασχόληση είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και άλλωστε έχει και αυξητική τάση. Και γνωρίζουμε επίσης ότι ήταν θερμοκήπιο η εποχική απασχόληση πάντα, θερμοκήπιο λέω της παράνομης εργασίας και όλης της μιζέριας που από αυτήν απορρέει. και ξέρουμε πολύ καλά ε, ότι στην χώρα μου, στην περιοχή του Ροζάτο, είχαμε ε, μια πολύ φρικτή ιστορία, την οποία πολύ συχνά αναφέρουμε όταν ε, μιλάμε για την εποχική απασχόληση. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απολύτως σωστό να πούμε ότι εάν έχουμε μια κοινωνικά σωστή αγορά, τότε δεν ε, θα ε, στρεβλώνεται και ο ανταγωνισμός. Σε μια αγορά η οποία υφίσταται το κοινωνικό ντάμπινγκ, οπωσδήποτε ε, ο ανταγωνισμός είναι απολύτως στρεβλωτικός. και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ε, ε, προχωρήσουμε όπως το κάναμε άλλωστε ε, και για τις ενδοεπιχειρησιακές αποσπάσεις και για τις μετακινήσεις εργαζομένων κλπ. Νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει κυρίως να αναφερθούν στο κείμενο το οποίο θα υποβληθεί στην ψήφο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Είναι μια σημαντική έκθεση αυτή για την Επιτροπή μας. Θα δώσω το λόγο, αφού είναι μαζί μας, στον ε, εισηγητή της Επιτροπής ε, Πολιτικών Λευθεριών, τον κύριο Κλοντ Μωράες. Thank you, Chair. And, um, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την πρόεδρο της Επιτροπής σας και τον κύριο Κοφεράτη για την πολύ καλή και στενή σχέση εργασίας που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Υπήρξα μέλος της Επιτροπής κατά το παρελθόν και γι' αυτό γνωρίζω πολύ καλά ότι και τα τρία ε, θέματα για τη λαθρομετανάστευση, η νέα άδεια, οδηγία, ICT και οι εποχιακοί εργαζόμενοι και τα τρία αυτά θέματα έχουν και ένα επίκεντρο που αφορά την αγορά εργασίας. Έχουμε το άρθρο 50, αλλά απαιτούνται στενές σχέσεις συνεργασίας γενικώ με τις, ε, μεταξύ της δικής σας επιτροπής και της δικής μας. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Κοφεράτη, αλλά να αναφέρω απλά κάποιους τομείς ε, επί των οποίων έχουμε κοινή αρμοδιότητα. Να αναφέρω επίσης ένα τομέα που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ίσως αυτό είναι το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσω. Δεχθήκαμε αυτά που περιλάμβανε η πρόταση τη Κομισιόν για το γεγονό ότι τα κράτη-μέλη ε, ελέγχουν πλήρως ε, και τους όγκους ε, και την έγκριση, την εισδοχή και πολύ σημαντικό θέμα ήταν αρχή της επικουρικότητας. Επίσης θέλει η Κομισιόν να γίνουν δοκιμές αγορά εργασίας και μετά ε, να αποφασίσει κατά πόσον θα δεχθεί μετανάστες. Αν δηλαδή οι θέσεις δεν μπορούν να πληρωθούν από τους ε, υπηκόους ε, είτε της χώρας είτε των χωρών της αυτό είναι πολύ σημαντικό και για σας φαντάζομαι. Τώρα, στα θέματα κοινή αρμοδιότητας, να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κοφεράτη, ότι εργαζόμαστε πολύ σκληρά σε ό,τι αφορά το τομεακό βεληνικές, την τομεακή εμβέλεια της πρότασης και συμφωνήσαμε να δούμε ε, και την γεωργία. και έναν άλλο τομέα και μετά ε, θα δούμε τι θα κάνουμε άλλους τομείς. Οι κοινωνικοί εταίροι επίσης πρέπει να συμφωνήσουν τι θα γίνει με, τον, ε, με την ε, γεωργία και τον άλλο τομέα που είναι ο βασικός, ο τουρισμός δηλαδή. Και την ε, γεωπονική. Το θέμα της εκμετάλλευσης των επιχειακών εργαζομένων που είπε και ο κύριος Κοφέρτη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οδηγία πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει πραγματική προσθέμενη αξία. Ορίσαμε τι θα πει αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης Είδαμε επίσης τα θέματα του υπερβολικού μισθώματος της εκμετάλλευσης των εποχιακών εργαζομένων. Καθώς επίσης και το κόστος το οποίο βαρύνει τον εργοδότη. Αλλάξαμε την πρόταση της Κομισιόν. Το κόστος έκδοσης βίζα και το κόστος ε, ταξιδίου θα το καταβάλει ο εργοδότης. Επίσης, Είπαμε ότι πρέπει να είναι αυστηρότεροι και πιο αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης και εισαγάγαμε και ένα τμήμα το οποίο μιλά για την πρόληψη της θυματοποίηση των εποχιακών εργαζομένων που έχουν υποβάλει καταγγελίες κατά το παρελθόν. Νομίζω λοιπόν ότι τις κοινέ μας αρμοδιότητες ε, τις έχουμε εξετάσει υπό το πνεύμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζετε και εσείς την επιτροπή σας στα θέματα της ισότιμης μεταχείρισης και όλα τα άλλα τα σημαντικά ζητήματα της έκθεσης. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είμαι μέλος Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, χαίρομαι που με έχετε για τη φιλοξενία, αλλά σίγουρα υπήρξε εξαιρετική συνεργασία. Και ίσως ε, δεν υπάρχει καλύτερη δυνατότητα να κάνουμε χρήση του άρθρου 50 από αυτό το τομέα. Η οδηγία για, τις εποχικές, ε, για τους σε σχέση με την αγορά εργασίας πραγματικά ε, επηρεάζει. Επηρεάζει πολύ την αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία που έχουμε και θα με ενδιαφέρει να ακούσω πάρα πολύ τις απόψεις των βουλευτών της Επιτροπής σας. Και μετά θα σας ενημερώσω και για τις αντιδράσεις ε, των μελών της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ, στην οποία μίλησε σήμερα ο κύριος Κοφεράτη, πρόεδρος. Πολύ ωραία. Βλέπω ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το πνεύμα του άνθρωπου 50 και αυτό με χαροποιεί η Ελίζα Σρέντερ είναι η πρώτη ομιλητρία. Ε, καταρχήν να πω ότι η θέση της ομάδας μας από την Τζιν θα εκτεθεί και παρουσιάζεται. Όμως μία ερώτηση έχω προς τον εισηγητή που με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Όταν λέτε ότι θέλετε τομείς να επιλέξετε που για αυτή την οδηγία θα εξεταστούν, τι θα γίνει σε σχέση με εκείνους τους εργαζόμενους που κατά κάποιο τρόπο προσέρχονται σε μια χώρα και δεν ανήκουν σε αυτούς τους τομείς αυτοί θα έχουν λιγότερα κοινωνικά δικαιώματα. Πώς θα διαμορφωθούν τα κοινωνικά τους δικαιώματα μέσα στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Δεν θα έχουμε πάλι μια διαφοροποίηση κοινωνικών δικαιωμάτων για αυτούς. Δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ε, monsieur le rapporteur, propose de, répondre à la fin. να στο τέλος. Jean Lambert. Thank you very much. Our, shadow on this is actually Emilia Turunen, who... Η Εμίλια είναι η αλλά δεν μπορούσα να είναι εδώ σήμερα και μου ζήτησε να πω εγώ εκ μέρους δύο-τρία λόγια. Εν γέννη, ε, συμφωνούμε με την προσέγγιση του εισηγητού στην Επιτροπή. Η ισότιμη μεταχείριση φυσικά είναι πολύ, ξέρετε, πολύ σημαντικό θέμα. Γνωρίζουμε από την άλλη βέβαια ότι αυτή η οδηγία δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα της εποχιακής εργασίας, γιατί ξέρουμε ότι υπήρξαν αντικείμενα εκμετάλλευσης, οι περισσότεροι των οποίων όμως ήταν υπηκόοι τρίτων, ε, μάλλον χωρών της Ένωσης που εργάζονταν σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν τη σημασία των προτάσεων του εισηγητή για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο και την ευθύνη των κρατών μετών και των αρμόδιων φορέων τους που θα πρέπει να φροντίσουν όποια νομοθεσία ισχύει να εφαρμόζεται στην πράξη. Γιατί μπορούμε να έχουμε την ισότητα μεταχείριση και την οδηγία, αλλά αυτός ο μηχανισμός επιβολής πρέπει να λειτουργεί ώστε να είναι αποτελεσματικό για όλους τους εποχιακούς εργαζομένους. για να έχουμε αξιοπρεπείς συνδικές εργασίας και ισότητα μεταχείριση. Επίσης το θέμα του μηχανισμού ε, υποβολή καταγγελιών που πρέπει να ενισχυθεί για το δικαίωμα προστασία των εποχιακών εργαζομένων μα χαροποιεί ιδιαίτερα. Και είναι καλό και για του ίδιου εργαζόμενου, αλλά και για τα συνδικάτα και για άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν εξ ονόματος των εποχιακών εργαζομένων. Και σε ό,τι αφορά την ιδιότητα του μέλου, ναι, και αυτό μπορούμε να το έχουμε ως δυνατότητα, αλλά είναι σημαντικό για ευάλωτου εργαζομένου. σε ό,τι αφορά το πεδίο, η τομιακή προσέγγιση ε, είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά γενικά μπορούμε να το στηρίξουμε και πρέπει να είναι ξεκάθαρη η περίοδος εργασίας που καλύπτουμε εδώ. Δεν θέλουμε να μην είναι σαφή τα όρια μεταξύ της απασχόλησης κάποιου ως εποχιακού εργαζομένου ή κάποιου που τον κρατά στη θέση του εργοδότης για μακρύτερο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως να του δίνει ένα άλλο καθεστώς. Η εξάμηνη περίοδος μέσα σε 12 μήνες και όχι η το ημερολογιακό έτος, αυτό είναι σημαντικό. Και η παροχή καταλήμματος είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε κάποια πρότυπα. Αλλά επαναλαμβάνω, έλεγχος και εποπτεία είναι σημαντικά. Γιατί πολλοί από του εργαζομένους ζουν σε απομακρυσμένε περιοχές και γι' αυτό άλλωστε είναι και πιο ευάλωτοι. Και εξού και τόσο σημαντικό να φροντίσουμε να του παρέχετε κατάλημα. Σε ό,τι αφορά το πρόσθετο κόστος, ότι θα πρέπει να πληρώσουν εργοδότες για τι θεωρίε διαβατήριου κτλ. Πρέπει να είναι σαφές ότι το κόστος αυτό θα είναι έξτρα πάνω από την αμοιβή. Δεν θα αφαιρείται από την αμοιβή. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και επίσης ό,τι αφορά τη σαφήνεια, τη μεγαλύτερη σαφήνεια για τις συλλογικές συμφωνίες, ποιες είναι εγκύρες και ποιες όχι, αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε. Και μάλλον θα υποβάλουμε μία-δύο τροπολογίες για να ενισχύσουμε τη σχετική διατύπωση και βέβαια παρότι θα κάνουμε τι τροπολογίε μας, νομίζουμε ότι η έκθεση πηγαίνει προ σωστή κατεύθυνση. Μάρια Χάρκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο σκιώδης μας δεν μπορεί να είναι εδώ και επομένως παίρνω εγώ την θέση του. Λέω λοιπόν ότι καλωσορίζουμε σαν πολιτική ομάδα την γνωμοδότηση αυτή. Όντως η εποχική απασχόληση είναι ένα σημαντικό ζήτημα ε, και πραγματικά η οικοδόμηση της ε, Ευρώπης είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει να πω ότι ε, η οδηγία της εποχικής απασχόλησης ε, είναι μέλος ε, των, του συνόλου των οδηγιών που διέπουν την αγορά και βεβαίως εμείς θέλουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Συμφωνούμε απολύτως με την ίση μεταχείριση. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι το κείμενο το οποίο θα εγκρίνουμε ε, οπωσδήποτε προβλέπει η συμμεταχείριση για όλους τους ε, εργαζόμενους. Ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες έτσι ώστε να μην έχουμε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη. Θα τα προσέξουμε τα σημεία αυτά. Γνωρίζουμε ότι οι εποχικά απασχολούμενοι αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, τους εκμεταλλεύονται και επομένως θα πρέπει και αυτοί να βεβαιωθούμε ότι θα χαίρουν των ιδίων ε, συνθήκων εργασίας με τους ε, υπηκόους των χωρών ε, της, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας υποδοχής φυσικά. Πιστεύουμε πάντως ότι γενικότερα η γνωμοδότηση πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει μεγάλη αντίθεση προς την οδηγία αυτή ε, από πλευράς πολλών κρατών μελών και γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Τέλος, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτούμε την προστιθέμενη αξία του κειμένου που ε, θα εγκρίνουμε. Αυτό το έγγραφο θα είναι καλό, θα είναι καλά νέα για την Ευρώπη εάν συμπεριληφθεί στο κείμενο αυτό ουσιαστικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Δεν τη θέλει. Πάρα πολύ ωραία. Θα ξαναδώσουμε λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας. Κύριε Κοφεράτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει στις ερωτήσεις τις οποίες μου υπευλήθησαν. Βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα αυτά ε, τα οποία είπαν. Ε, το πνεύμα των παρεμβάσεών τους ε, πραγματικά δείχνει ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία και έχουν διάθεση συνεργασίας. Στην κυρία Σρέτερ να πω ότι στόχος είναι να υπάρχει μία και μόνη αγορά εργασίας και όχι να δημιουργήσουμε έστω και άθελά μας διαφοροποίησης. Όταν θα απομονωθούν οι τομεί δραστηριότητας δεν θα υπάρχουν άλλοι εποχικοί απασχολούμενοι. Επίσης, η διατύπωση ε, βάσει της οποίας ορίζεται τι, τι περιλαμβάνει η εποχική απασχόληση και ο εποχικά απασχολούμενος ε, είναι κάτι που μας απασχόλησε πολύ και το συζητήσαμε. Επιλέξαμε την πιο αποτελεσματική κατά την απόψή μου ε, δυνατότητα, δηλαδή να αναφέρουμε εργασίες οι οποίες επηρεάζονται από τον κύκλο των εποχών. Γι' αυτό ακριβώς καταλήξαμε σε αυτές τις τρεις που είναι δύο στην ουσία. Ε, δηλαδή γεωργική, γεωργικές εργασίες, λαχανικά και τουρισμό, Οι δύο πρώτοι μπορεί να θεωρηθεί ένα τομέα δραστηριότητας. Οτιδήποτε πλην αυτών των τομέων και των δραστηριοτήτων δεν μπορούν να θεωρηθούν εποχική απασχόληση. Τα, οι υπόλοιπε δραστηριότητες μπορούν να οριστούν ως προσωρινές εργασίες και όχι ως εποχικές. η κυρία Λάμπερτ έκανε μία ε, αναφορά στα χρονικά διαστήματα. Έξι μήνες θεωρούμε ότι είναι ένας ικανός χρόνος για ε, μια εποχική δραστηριότητα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δικαιολογηθεί μεγαλύτερη περίοδος, έστω και αν σε ορισμένες χώρες με εποχική απασχόληση εννοούμε ε, ε, απασχόληση ε, σε πιο μεγάλο διάστημα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με το εξάμεινο βασιζόμενοι βεβαίως στο 12μηνο σύστημα το οποίο έχουμε, γιατί ε, ξέρουμε ότι βάσει του ηλιακού ε, συστήματος ορίζονται οι περίοδοι της ε, γεωργίας. Ε, και εκεί δεν περνάμε από τη μία χρονιά στην άλλη. Ο τουρισμός μπορεί να ε, ξεπεράσει το ημερολογιακό έτος, δηλαδή μπορεί ο χειμερινός τουρισμός να ξεκινήσει στον προηγούμενο χρόνο και να τελειώσει στον επόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτήν την ε, στοιχειώδη διάρθρωση που υπάρχει στους τομείς δραστηριοτήτων που απομονώσαμε, αυτούς τους τρεις τομείς. Πολλές φορές είπαμε μεταξύ μας ότι θα πρέπει να ενοποιήσουμε την αγορά εργασίας και ότι θα πρέπει για ίδια απασχόληση να υπάρχει ίδια αμοιβή, για ίδια απασχόληση ίδιες συνθήκες. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός ευαισθησίας για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι οι συνθήκες που διέπουν την εποχική απασχόληση είναι εξαιρετικά στρεβλωμένες αλλά ότι παρόλα αυτά η γενικότερη τάση είναι μία στάση ευαισθητοποίησης απέναντι στο θέμα που θα μας επιτρέψει νομίζω να κάνουμε αυτά τα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση που όλοι επιθυμούμε. Δηλαδή ίση μεταχείριση, καμία διάκριση έστω και άθελά μας. Βεβαίως θα υπάρξουν και οι τροπολογίες επί των οποίων θα συζητήσουμε πάλι. Πάντως σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που κάνατε και κυρίως για το πνεύμα με, τον οποίο, με το οποίο αντιμετωπίσετε το κείμενο αντικείμενό μου. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τώρα θα φτάσουμε ε, στα πιο δύσκολα, 22 Ιουνίου έχει, έχει οριστεί η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ξέρω ότι είναι μικρό το, το διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Παρακαλώ τους συναδέλφου λοιπόν ε, να υποβάλουν τροπολογίες μέχρι τι 22. Ε, σημείο 23 λοιπόν, η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο και μιλάμε για όλα τα τμήματα, επ' αυτόν πρέπει να υποβάλω γνωμοδότηση. Ξέρετε ότι ε, μπερδεύτηκαν λίγο τα πράγματα με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, και προσπαθούμε να φτάσουμε σε μία ε, σύμφωνη γνώμη όσον αφορά το προϋπολογισμό 2012. Ε, Αυτός θα μας απασχολήσει στην επόμενη μήνυ ολομέλεια. Και η γνωμοδότηση την οποία συζητούμε σήμερα αφορά την απάντησή μας ακριβώς για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012. Η Επιτροπή έχει υποβάλει το σχέδιο προπολογισμού το, το τέλη Απριλίου και περιμένουμε άλλωστε και τώρα και τη θέση του Συμβουλίου και βάσει της θέσεως του Συμβουλίου ε, θα πρέπει να εργαστούμε και να υποβάλουμε τις τροπολογίες μας. Το έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας, ε, αν επαναλαμβάνω όλα τα μελήματα τα οποία εμείς έχουμε εκφράσει στη διάρκεια του τριμερού στη διαλόγου, και μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο ε, στάδιο, δηλαδή όπου θα μιλάμε πλέον για συγκεκριμένα στοιχεία με συγκεκριμένους αριθμούς sur le fond... και υπολογίζουμε ότι αυτό θα γίνει περί τα τέλη του καλοκαιριού. Επί της ουσίας όμως δεν έχουμε καμία τροποποίηση όσον αφορά τις προτεραιότητες τις οποίες από κοινού και μέσα από κοινή συμφωνία αποφασίσαμε. Λαμβάνοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία υπόψη σας προτείνω να θεωρήσετε ότι αυτή η γνωμοδότηση δεν χρειάζεται έτσι μεγάλη ε, συζήτηση και μακροσκελής παρεμβάσεις. Συμφωνούν οι συνάδελφοι. Συμφωνούν όλοι. Όχι, η κυρία Άρκιν θέλει να μιλήσει. Για αυτό το σημείο το οποίο συζητάμε δεν έχω μίζωνα θέματα να παρουσιάσω. Μια και έχω τον λόγο θα είμαι πολύ σύντομη όμως. Δύο ερωτήσεις έχω που θα ήθελα να θέσω. Σύμφωνο με τα περισσότερα τα οποία αναφέρθηκαν, με όλα τα όσα είπατε σε σχέση με την νέα κατηγορία για ενδιάμεσες ε, περιφέρειες. Η ομάδα του Άλντε είναι κατά και η ερώτησή μου θα ήταν ποια είναι η πρόσθετη αξία να υπάρχουν ενδιάμεσες περιφέρειες. Τι προσφέρει αυτό επιπρόσθετα. Νομίζω αυτή είναι η μόνη ερώτηση που έχω, αν είναι δυνατόν να απαντηθεί. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ συνάδελφοι, θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το είχαμε δει όταν εξετάσαμε και το σχέδιο γνωμοδότησής. Δεν μπορώ να μπω στην ουσία τη συζήτηση. Θα σας πρότεινα όμως να επανέλθουμε όταν θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. γιατί είναι κρίμα να χάσουμε τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε με τον Επίτροπο παρόντα. Λοιπόν, το έγγραφο του Συμβουλίου θα μας ε, δοθεί μετά τη συνάντηση της Κορεπέρ τον Ιούλιο και θα εγκριθεί οριστικά την 21 η εβδομάδα και με βάση αυτό το έγγραφο του Συμβουλίου που τροποποιεί τη θέση της Κομισιόν μπορείτε και εσείς να καταθέσετε μέχρι τις 24 Αυγούστου τις δικές σας τροπολογίες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της Μέσης Διάταξης και με χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας ε, τον Επίτροπο, τον Επίτροπό μας. Σας ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε αλλά μιλούσαμε για τους εποχιακούς εργαζομένους, ένα πλοκό θέμα όπως γνωρίζετε. Δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ξέρω ότι θέλετε να μιλήσετε και γενικά για το πρόγραμμα εργασίας σας, αλλά ξέρετε για μας η επικαιρότητα ε, βασίζεται ουσιαστικά στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας. Το περίφημο πρόγραμμα των συστάσεων για τα εθνικά προγράμματα, τις ειδικέ δηλαδή κατά χώρα συστάσεις. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά να είμαι ενώπιον σας και να συζητώ σημαντικά θέματα μαζί σας. Ελπίζω ότι το γεγονός ότι έπρεπε να περιμένω εκτός δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει λιγότερος χρόνος για τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα μπορούμε να είμαστε ουσιώδεις και στη συζήτηση όπως πάντα. Υπάρχουν κάποια πραγματικά σημαντικά θέματα για αυτή τη συζήτηση και όταν για πρώτη φορά είχαμε την προοπτική αυτής τη συζήτησης είχαμε και το πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2012 βρισκόμαστε σε μια πρώιμη φάση αρκετά νωρίς παρόλα αυτά θεώρησα ότι καλό θα ήταν τις προτάσεις μου να τις, ε, σας, παρουσίαζα σε αυτή την πρώιμη φάση και να έχω τις αντιδράσεις σας, τις τοποθετήσεις σας ε, προτού τεθούν αυτές οι προτάσεις στο Συλλογικό Σώμα των Επιτρόπων. Το άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό το οποίο προανέφερε η κυρία Πρόεδρος. Οι πρώτες συστάσεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ουσιαστικά που στοχεύουν να διασφαλίσουν τον συντονισμό οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών και αν μου επιτρέψετε θα ξεκινήσω με το δεύτερο θέμα και μετά θα επιστρέψω στο πρώτο. Τώρα, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, η στρατηγική της Ευρώπης 2020 είναι αυτή στρατηγική για την αηφορία στην ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, συμφωνήθηκε. Τώρα θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 2020 ε, και των κυριότερων πρωτοβουλειών. Αυτά που υιοθετήθηκαν στις 7 Ιουνίου αφορούν αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα για κάθε κράτος μέλος που θεωρώ ότι είναι τα πιο ουσιώδη βράχη πρόθεσμα για να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό για την ανταγωνιστικότητα και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης αντιμετωπίζοντας όμως ταυτόχρονα και τις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα προβλέπουμε και τις μακροπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ε, δράσεις ε, για την αναγκαία ανάπτυξη και τις αναγκαίες ε, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και οι συγκεκριμένες συστάσεις για τις χώρες για να υποστηριχθούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την δημοσιονομική παγίωση και πειθαρχία μέχρι και την, ε, τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας. Οι συστάσεις μας βασίζονται σε δύο ουσιώδεις νομικές βάσεις το άρθρο 121.2 και το 48.4 που πρέπει να διασφαλίζεται η ολοκληρωμένη εφαρμογή τους. Είναι σαφές ότι είναι διαφορετικές οι προκλήσεις μεταξύ κρατών μελών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που αφορά συγκεκριμένες ιδιομορφίες των κρατών μελών επικεντρωνόμενοι σε συγκεκριμένες προκλήσεις όπως ε, για τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων π.χ. Την, ε, ε, τα διαθωτικά θέματα όσον αφορά την απασχόληση, μείωση του κατακαιρματισμού της αγοράς εργασίας και αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, βελτίωση των συστημάτων παιδείας και εκπαίδευσης και διασφαλίζοντας ότι θα μπορούν ανάλογα με την αύξηση της παραγωγικότητάς τους να αντιμετωπιστούν οι ε, περιφέρειες και κάθε ένας. Έτσι θα πρέπει οι αποτελεσματικές ε, αυτές ε, απαντήσεις να προσπαθήσουμε να εξευρεθούν μέσα από αυτό το πλέγμα. Υπάρχει μία διασύνδεση μεταξύ των συστάσεων και της ετήσιας επισκόπησης όσον αφορά την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, της βελτίωσης ε, της περίθαψης και φροντίδας των παιδιών και πολλών άλλων θεμάτων, επικεντρωνόμενοι και όσον αφορά τις ανάγκες των συστημάτων εκπαίδευσης, όσον αφορά την αγορά εργασίας κτλ δίνοντας κίνητρα τώρα για την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας το συνταξιοδοτικό όριο και βελτιώνοντας την προσπελασιμότητα για την φροντίδα παιδιών. Είναι κύρια προτεραιότητα σε πολλά κράτη-μέλη για το άμεσο μέλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό με τις δημογραφικές αλλαγές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Η οικονομική κρίση αύξησε την διαθροτική ανεργία και έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ευάλωτων ομάδων. Είναι ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και μάλιστα κατεπηγόντως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι ζωτική σημασία να βελτιώσουμε τις ε, διαδικασίες στην ε, αγορά μειώνοντας το φορολογικό βάρος ε, και την επιβάρυνση όσον αφορά τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενους. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η δραστηριοποίηση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, καθώς επίσης και η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης με στοχοθέτηση ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πάλι. Πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε. Να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βελτιώσουμε τις προοπτικές για τους νέους, να μειώσουμε τα επίπεδα ανεργίας των νέων και την, το φαινόμενο των νέων που εγκαταλείπουν τα σχολεία υπερβολικά νωρίς πρόημα χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδέ τους και η διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και δυνατότητας κατάρτισης ώστε να βρουν απασχόληση οι νέοι στη συνέχεια πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να ε, δώσουμε κίνητρα για την ε, οικονομική ανάπτυξη και αυτά να, να λάβουν πάντα υπόψη, να λαμβάνουν υπόψη και την παραγωγικότητα. Σε κάποιες χώρες θα πρέπει να υπάρξουν ίσως και αλλαγές στα συστήματα διαπραγμάτευσης των ε, συλλογικών συμβάσεων και μισθολογικών ε, όρων για την απασχόληση μεταξύ των συμβαλωμένων μέρων. Πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων, ιδιαίτερα μεταξύ της ανάγκης για δημοσιονομική πειθαρχία και εξυγίανση και την ανάγκη του να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές συνιστώσεις σε σχέση με κάποιες δράσεις. Συστάσεις για τις συντάξεις είναι ένα καλό παράδειγμα προς αυτά ενώ αρχικά έχουν προσεγγιστεί για να βελτιωθεί η αηφορία των δημοσιονομικών έχουν ουσιώδη ρόλο για κάποια κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης μείωσης ή συρρήκνωσης του εργατικού δυναμικού. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνεται υπόψη, λαμβάνονται υπόψη τα μελήματα και οι ανησυχίες ιδιαίτερα για εκείνες τις χώρες όπου το επίπεδο φτώχειας για τους ε, ηλικιωμένους, ιδιαίτερα για τις ε, ηλικιωμένες γυναίκες είναι πολύ υψηλό. Θέματα φύλου επίσης ε, καλύπτονται, λαμβάνοντας υπόψη την χαμηλή συμμετοχή πολλές φορές των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το πακέτο αυτού του, της 7ης Ιουνίου θα το συζητήσω με τα κράτη-μέλη αύριο στο Συμβούλιο και θα δούμε αυτά από κοινού. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι σαφές για μένα ότι το 2012 το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να επικεντρώνεται στις ε, πρωτοβουλίες ναυαρχίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στρατηγική του 2020. Προτίθεμαι να αναλάβω ε, πρωτοβουλίες σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες ως τομείς. Πρώτον, σαν συνέχεια τη ατζέντα για τι νέε δεξιότητε και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ένα ολόκληρο πακέτο για την απασχόληση θα παρουσιαστεί με διαφορετικέ πρωτοβουλίε για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, δεξιότητε, διακυβέρνηση, βελτιώνοντα το δίκτυο για του νέου στην Ευρώπη, δημιουργώντα ένα νέο κίνητρο για την flex security, την ασφάλεια και ελαστικότητα. Η αρχή τη ασφάλεια και ελαστικότητα, flex security, που συμφωνήθηκε το 2007, είναι μέσα σε ένα ε, καλά ισορροπημένο ισορροπημένο αναλογικό πλαίσιο όμως παρόλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπήρξε αύξηση της ανεργίας, μεγαλύτερος κατακαιρματισμός στην αγορά εργασίας και αντιμετωπίζουμε και πιο στενά δημοσιονομικά όρια. Πρέπει να έχουμε ελαστικότητα, να δοθούν κίνητρα για να υπάρχει και ελαστικότητα και ασφάλεια, ώστε να μπορέσουμε αυτή την περίοδο να την γεφυροποιήσουμε, να την καλύψουμε καλύτερα εξετάζουμε και διερευνούμε νέε δυνατότητε για την μεταρρύθμιση των αγορών εργασία με του κοινωνικού εταίρου και με τα κράτη-μέλη ω εταίρου. Αποκινούμε αυτή την, με αυτό το ερωτηματολόγιο και την επισκόπηση υποβάλαμε διαφορετικές προτάσεις για τη μεγαλύτερη χρήση της εσωτερικής ελαστικότητας και την επέκταση των ε, ε, ε, ευεργετημάτων σε εκείνους ε, που ακόμα μπορεί και να μην έχουν ε, και απασχόληση. Για παράδειγμα, το θέμα των συμβάσεων έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις. Αυτό δείχνει την ανάγκη να, υπάρξουν, να υπάρξει εμβάθυνση στις συζητήσεις οι εμπλεκόμενοι να δουν καλύτερα τα θέματα της ελαστικότητας και ασφάλειας, ε, flex security, πράγμα που πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2012 θα υποβληθούν εξειδικευμένες συγκεκριμένες προτάσεις με αποτέλεσμα αυτή τη διάσκεψη, τα συμπεράσματα αυτής της διάσκεψης, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της πρώτης φάσης της ελαστικότητας, δηλαδή της περίοδου 2007-2010. Σε αυτή τη φάση φυσικά είναι υπερβολικά πρόημο να σχολιάσουμε και να προβλέψουμε κάποια τελική έκβαση τελεσίδικα. Επιπλέον, ως μέρος της πρωτοβουλίας ε, οι νέοι ε, σε κίνηση, οι νέοι κινητοποιούνται, youth in movement, έχουμε υπόψη να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, μπορούν να υπάρχουν και υποτροφίες και υποστήριξη για τους νέους και να καλύψουμε το κενό μεταξύ θεωρητικών γνώσεων και των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται και χρειάζονται στους χώρους εργασίας. Πρέπει όμως να αποφύγουμε καταστάσεις όπου θα αποτελέσουν αντικείμενο κατάχρησης ε, αυτές ε, οι δυνατότητες ε, και να υπάρχει και η δυνατότητα μαθητείας και περίοδου μαθητείας για την απόκτηση γνώσεων και απόκτηση θέσεων εργασίας. Με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2010 για την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας λαμβάνεται αυτό υπόψη, καθώς επίσης και το θέμα της έκθεσης της κυρίας Τούρουνεν. Αξιότιμα μέλη, ένας από τους κυριότερους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής είναι να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερης ποιότητας αναβαθμισμένες θέσεις απασχόλησης. Αυτό δεν θα μπορεί να είναι δυνατόν αν δεν διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Υποστηρίζοντας αυτό το στόχο, κατά τα τέλη του 2012 θα υποβληθεί μια νέα πρόταση όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία ε, στον στο χώρο εργασίας ε, μέχρι σε ένα πολιετές πλαίσιο. Θα έχουμε πρωτοβουλίες σε δύο άξονες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Πρώτον, μία πρόταση θα υποβάλουμε για τις μειοσκελετικές ε, ε, παθήσεις κατά τη διάρκεια του 2011 ήδη. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτό το θέμα πρέπει σε εθνικό επίπεδο να καλυφθεί, να αντιμετωπιστεί και μια νέα πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και αυτή την πτυχή. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι ενώ βλέπουμε ότι και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό επίπεδο έχουν αναλυφθεί πρωτοβουλίες, παρόλα αυτά εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε θα πρέπει σε σχέση με τις μυοσκελετικές ε, παθήσεις να πούμε ότι αφορούν 61% όλων των συνεπαγωμένων ε, προβλημάτων σε σχέση με την υγεία και τις ε, περιόδους ασθένειας των εργαζομένων. Θα αξιολογηθούν όλοι οι παράγοντες κινδύνου στους χώρους της εργασίας για να διασφαλίσουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ένα ολοκληρωμένο και απλουστευμένο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την υγεία που θα είναι πιο αποτελεσματικό και πιο εύκολο να εφαρμόζεται. Δεύτερον, προτίθεμαι να υποβάλω μια πρωτοβουλία που θα προστατεύει τους εργαζομένους όσον αφορά την έκθεσή τους σε καπνό στην εργασία τους. Και σε σχέση με την φάση αυτή της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους που θα ξεκινήσει εφέτος, μια μελέτη βρίσκεται υπό για να υποστηριχθεί η δεύτερη αυτή φάση ε, συζήτησης και εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων. Ω μέρο αυτή τη πρωτοβουλία μπορεί να υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομοθετική πρωτοβουλία και οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να ήθελαν να υπησέλθουν σε διαπραγματεύσει. Αν γίνει αυτό και στεφθεί με επιτυχία μια τέτοια συμφωνία, τότε θα οδηγηθεί σε μια οδηγία του Συμβουλίου με βάση μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για να ευδοκιμήσουν αυτοί οι στόχοι. Θα ήθελα να δραχθώ αυτή τη ευκαιρία να ενημερώσω ότι πριν από δύο ημέρε υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πρόταση για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παρακολουθήσατε ως θέμα εκ του σύνεγγυς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή εσεί. Αφορά τις αρχές της καλύτερης ε, βελτιωμένης νομοθεσίας διασφαλίζοντας ένα συγκεκριμένο βαθμό ε, ελαστικότητας και αναλογικότητας ε, καθώς επίσης και ιατρικής εποπτείας και παρακολούθησης. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα τα συμφέροντα της υγείας, την υγεία των εργαζομένων που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά παιδεία. Ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί κατά τα τέλη της του επόμενου έτους ε, η πρόταση αυτή και από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, σήμερα σχεδόν 23 εκατομμύρια πολίτες είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνω από 113 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται στο κατόφλι της ε, φτώχειας ή και του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πραγματικά ανησυχητικά αυτά τα μεγέθη. Ωστόσο ακόμα πιο ανησυχητικά είναι η, τα, είναι ανησυχητική αριθμή των παιδιών που ζουν στην φτώχεια και αποκλεισμό περισσότερο από των ενηλίκων. Επιπρόσθετα ξέρουμε ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα αυτά τα παιδιά. Αυτά που ζουν με έναν και μόνο γονέα ή ζουν σε ένα νοικοκυριό που είναι ε, άνεργος ο γονιός και η φτώχεια πραγματικά είναι η μεγαλύτερη απειλή. Πρέπει μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να υποβάλουμε μια πρόταση για την αντιμετώπιση της ε, κατάστασης αυτής των παιδιών. Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία κοινών αρχών και πλαισίων ώστε να έχουμε μια δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βέλτιστες προδιαγραφές. Καθορισμός κοινών αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για δράση σε τρεις τομείς, σε τρεις άξονες. Πρώτον, υποστήριξη οικογενειών για παράδειγμα, σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και υποστήριξη εισοδημάτων, επιδομάτων δηλαδή. Δεύτερον, στην περίθαλψη και φροντίδα παιδιών, στη στέγαση και στις κοινωνικές υπηρεσίες, υποστήριξη πάλι και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, ένταξη στην κοινωνία. Φυσικά, τα παιδιά δεν είναι η μόνη ομάδα που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι νέοι, οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι, οι ηλικιωμένοι και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Τον προηγούμενο μήνα είχε γίνει ένα σημαντικό βήμα για την ένταξη των Ρωμά των Τσιγκάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για στρατηγικές για τη μειονότητα αυτή για τους ε, Τσιγκάνους. Είναι ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα ότι από πλευρά μα δεν θα δεχτούμε εμεί την τον κοινωνικό αποκλεισμό των τσιγκάνων, των Ρωμά. Είναι σαφέ ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη είναι τα πρώτα κυρίαρχα για τον καθορισμό και την κατάρτιση στρατηγικών όσον αφορά την ένταξη των τσιγκάνων. Παρόλα αυτά, ωστόσο, τούτων λεχθέντων πιστεύω στεναρά ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό έχει ένα σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει. Το πλαίσιο υπογραμμίζει την πρόσθετη αξία συντονισμένων δράσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μα δώσει την ευκαιρία να ε, ε, συγχωνέσουμε και να συγκλίνουμε με τις πολιτικές μας, ε, τις στρατηγικές μας εκείνες για την ε, ένταξη των Ρωμά και την κινητοποίηση των κονδυλίων. Το Συμβούλιο έχει ήδη υιοθετήσει αυτή την ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των τσιγκάνων και βασίζομαι στην υποστήριξη της Ευρωβουλής, ιδιαίτερα της δικής σας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, για να υπάρξουν αλλαγές χειροπιαστές επιτόπου σε σχέση με τους τσιγκάνους. Κυρίες και κύριοι, η ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και την απασχόληση προσανατολίζεται σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε για χαμηλές εκπομπές ρήπων, διοξιδίου του άνθρακα και προστασία του περιβάλλοντος. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν διατυπώσει αυτά τα αιτήματα. Το 2011 μια δημόσια συζήτηση θα ε, πάρει το εναρκτήριο λάκτισμα ώστε να βρεθούν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας τους στον πυρήνα αυτών των στρατηγικών θα αναζητηθούν τρόποι να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα των πολιτικών και στρατηγικών για την αηφορία στην ανάπτυξη. Επίσης θα δούμε πώς μπορεί να διευκολυνθεί η μετάβαση και στην ε, ε, τοπική και περιφερειακή ε, αηφόρο οικονομία καθώς επίσης ε, και την, ε, πιο τη μεγαλύτερη απόδοση. Θα δούμε και την μετάβαση στην οικονομική, θέματα που αφορούν την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική καινοτομία, το πρασίνισμα της οικονομίας και της κοινωνίας και τις αλλαγές που συνεπάγονται όλα αυτά. Στοχεύω να υποβάλω μια ανακοίνωση το 2012 που θα σκιαγραφεί συγκεκριμένες και εξειδικευμένες δράσεις σε αυτούς τους τομείς. Λοιπόν, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η Ευρώπη, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Από το 2012 η ηλικία, θα, ε, το, εργατικό δυναμικό θα αρχίσει να συρρυκνώνεται, ενώ θα αυξάνεται η ηλικία των εργαζομένων και μάλιστα ε, των ηλικιωμένων κατά 2 εκατομμύρια ετήσια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξελίξεις όσον αφορά τη δημοσιονομική συνιστόσα. Το 2012 θα είναι ένα σημαντικό έτος ως προς αυτά. Πρώτον, το 2012 ήδη έχει προκαθοριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος για την δραστήρια γύρανση καλωσορίζω τη συμμετοχή με του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξειδικευμένε δράσεις. Δεύτερον, θέλει να δραχθεί τη ευκαιρία για τη μοναδική συγκυρία για το ευρωπαϊκό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζοντα μια ανακοίνωση με μηνύματα για την πολιτική όσον αφορά την υπεργύρανση και την ενεργό γύρανση και την συμμετοχή αυτών των πολιτών στο κοινωνικό ε, γίγνεσθε. Τρίτον, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της προστασίας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, εκείνων που αλλάζουν και θέση εργασίας. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την τροχοπέδη που υφίσταται αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και να άρουμε τα προσκόμματα όσον αφορά ε, την συνταξιοδοτική αυτή ε, ε, κάλυψη των εργαζομένων. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση της κατάρτισης και της διατύπωσης των προτάσεων για αυτή την πολιετή περίοδο. Και αυτό είναι το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να καλύψω στην εισαγωγική μου αυτή παρέμβαση. Θα ήθελα να δραχθώ λοιπόν της ευκαιρίας και να υπογραμμίσω έτσι ένα άλλο ζήτημα. Θέματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν κέρια σημασία σε σχέση με τις συζητήσεις που διεξάγονται σήμερα. Μια αξιόπιστη πρόταση από πλευράς μας πρέπει να αντανακλά τις αλλαγές ε, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες και θα πρέπει να προσφέρει και λύσεις για αυτά τα προβλήματα. Η ανεργία είναι ο υπαριθμό ένα ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να ενεργοποιηθούμε με πιο δραστήριο τρόπο επ' αυτού. Πλήρης ευθυγράμμιση με, τη στρατηγική, με τους στόχους της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020. Θα πρέπει περαιτέρω να επενδύσουμε στους πολίτες. Οι κοινωνικές αυτές επενδύσεις είναι σημαντικότατες για τη μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα, για την οικονομική και κοινωνική μας συνοχή και την αξιοπιστία της στρατηγικής μας για το 2020. Γι' αυτό προτείνουμε μια πρωτοβουλία για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, βασιζόμενη στην απασχόληση, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις προοπτικές για το μέλλον. Και κατά αυτή την έννοια το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πολύ σημαντικό και παίζει σημαντικό ε, ρόλο και επομένως θα πρέπει ε, να ενισχυθεί ο ρόλος του. Βεβαίως ε, θα πρέπει να δοθεί ε, μέσω του Ταμείου δυνατότητα κυρίως ε, στις πιο φτωχές χώρες να δώσουν μια νέα όθηση στο δυναμικό της απασχόλησης. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες συστάσεις τις οποίες ανέφερα και προηγουμένως και όλες οι προτάσεις μας συνδέονται με την ορθή επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. Βεβαίως θέλουμε και συνέχιση επικοδομητικής πολιτικού διαλόγου μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Και φυσικά εγώ θέλω να συνεχίσω να δουλεύω στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα και με την Επιτροπή Απασχόλησης ειδικότερα, όχι μόνο μέχρι το 12 αλλά και πέρα από αυτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για αυτά τα τόσο σημαντικά και εξαντλητικά ε, που μας είπατε. Δυστυχώς ε, θα πρέπει να περιορίσω λίγο στα δύο λεπτά τον χρόνο παρέμβασης. Ο κύριος Αλέξανδρος Θέρκας και μετά... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίγα είναι τα δύο λεπτά. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας ε, ευχαριστήσω κύριε Πίτροπε και μετά να σας ε, λυπήσω. Λοιπόν, ε, καταρχάς πριν από ένα χρόνο κύριε Πίτροπε ξεκινήσαμε να συζητούμε τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και σήμερα μας παρουσιάσατε το έγγραφο εργασίας. Και το έγγραφο για τις 7, ε, αλλά κάποια στιγμή θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά και για, την, ε, για το πρόγραμμα εργασίας. Η ανεργία πράγματι είναι η βασικότερη ανησυχία για τους Ευρωπαίους πολίτες, για να μην πω μια τραγωδία, ένα δράμα που βιώνει η Ευρώπη. Ανησυχεί πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφού διάβασα τι συστάσει προ τα κράτη-μέλη, νομίζω ότι η ύψιστη ανησυχία τη Κομισιόν δεν είναι η ανεργία, αλλά η δημοσιονομική εξυγένση πραγματικά εντελώς ε, ανισόρροπα βλέπετε τα πράγματα. Ε, έχετε προγράμματα που μιλούν για περικοπές, περιστολές, ε, που περιστέλουν όμως πράγματα πολύ σημαντικά για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και σε μια περίοδο δραματικής κατάστασης για τα δημοσιοοικονομικά, τα χρονοδιαγράμματα είναι αδύνατο να εκπληρωθούν ε, και η ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση και οι επενδύσεις ε, πρέπει να ε, αυξηθούν, όχι να μειωθούν. Μαμά, πώς μας λέτε λοιπόν ότι σας ενδιαφέρει η ανεργία, σας ενδιαφέρει η δημοσιονομική εξυγίανση και στην ανακοίνωση τύπου είπατε ότι υπάρχει μια βαθιά τεχνική μελέτη που δίνει απαντήσεις και κάνει προτάσεις πολιτική φύσεως πρέπει να είναι η μελέτη που θα γίνει, κύριε Επίτροπε, σε αυτή τη δραματική περίοδο που βιώνει η Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι εσείς προσωπικά έχετε μια μεγάλη πολιτική ε, ευαισθησία. Δεν πρέπει να βασίσετε τόσο σε αυτά που σας λένε οι ανώτεροι υπάλληλοι της ε, Κομισιόν. Μειώνουμε το κοινωνικό κόστος, τις κοινωνικές δαπάνες ε, χωρίς να πλήξουμε τον πληθυσμό που σφίγγει το ζωνάρι περισσότερο, που ε, περικόπτουν ε, τα επιδόματά του, οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται τελικά οι δημόσιε υπηρεσίε, οι κοινοφελεί υπηρεσίες, η υγεία, οι υγειονομικέ υπηρεσίες πλήττονται. Λυπούμε πραγματικά που θα το πω κύριε Επιτροπε, αλλά η σοσιαλιστική ομάδα έχει ε, πραγματικά διακατέχεται από βαθιά απογοήτευση. Αναποτελεσματικά άδικα είναι αυτά τα μέτρα και τελικά θα επιδεινώσουν το πρόβλημα και δεν θα το επιλύσουν. Ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά κάνει να αγωνιά εκατομμύρια κόσμο. Φρεντερίκ Νταρντέν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα επικεντρωθώ μονάχα στις, στις τάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η παρέμβασή σας η εισαγωγική είναι ενδιαφέρουσα κατά κάποιο τρόπο ή από κάποιες απόψεις και αρκετά εξαντλητική. Αλλά όπως ε, είπε προηγουμένως ε, και ο συντονιστής της ομάδας μου, με κεντρίζουν πολλά από αυτά που είπατε. Ε, οι συστάσεις στα πλαίσια της διακυβέρνησης μερικές φορές και μάλλον λίγο περισσότερο από μερικές, αρκετές φορές, μου φαίνονται λίγο περίεργες και αμφιλεγόμενες λέμε να προωθήσουμε μια Ευρώπη έξυπνη ε, που θα ε, ε, έχει κοινωνική ολοκλήρωση κτλ. Ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι δεν θα υπάρχει απαραίτητη κοινωνική κάλυψη και κοινωνική προστασία χωρίς γραμμές του προϋπολογισμού ενισχυμένες όσον αφορά και τα κράτη και την ε, Ένωση. Δεν μπορώ να καταλάβω ε, τι μπορώ να πω και τι προτάσεις μπορώ να κάνω για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας που παρόλα αυτά από ό,τι λέτε είναι μία από τις ε, προτεραιότητές σας γιατί δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί χωρίς το συμπληρωματικό προϋπολογισμό. Επίσης δεν σέβεστε κάνοντας κάποιες προτάσεις μερικούς από τους κοινωνικούς εταίρους όταν ας πούμε συστήνεται ότι ο τρόπος ο τρόπος ε, μισθοδοσίας, μάλλον καθορισμού των μισθών του Βελγίου ε, μέσω της αυτόματης συμπεριφερικής αναπροσαρμογής ε, στο Βέλγιο θα πρέπει να αλλάξει, δεν σέβεστε τον τρόπο υπολογισμού. Γνωρίζω βεβαίως ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Στη συζήτηση για την έκθεση ε, για την πράσινη ε, βίβλο εμείς καταφέραμε να διαγράψουμε ε, την ηλικία συνταξιοδότηση που ήταν σχετιζόμενη με το προσδόκιμο ζωής αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μας δημιουργούν πρόβλημα. Ελίζαμπετ Λίβερ και μετά η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ πολύ. Οι συστάσεις είναι ε, αρκετά τα ικανοποιητικές. Ε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα κράτη-μέλη ε, θα έπρεπε να έχουν λίγο περισσότερο χρόνο για να το μελετήσουν πριν την τελική του μορφή. Εν πάση περιπτώσει, ε, χαίρομαι που ε, ολοκληρώθηκε η οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά ε, ε, ε πεδία και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το έχουμε δουλέψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που ολοκληρώθηκε η δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε λίγο και γι' αυτό. Um, uh, όσον αφορά την οδηγία για τις μυοσκελετικές παθήσεις. Ε, γνωρίζω βεβαίως ε, ότι ε, αυτή η οδηγία μαζί με την οδηγία για τις χειρονακτικές εργασίες έχουν συντονισμένα προωθηθεί. Όμως θέλω να μου πείτε, θα κάνετε κάτι καινούργιο ή θα βασιστείτε στην υπάρχουσα νομοθεσία. Επίσης, κάπνισμα και παθητικό κάπνισμα δεν έχω τα στοιχεία πόσες χώρες μέλη δηλαδή έχουν ε, έχουν ενσωματώσει την νομοθεσία για τον καπνό και δεν έχω και στοιχεία τι ακριβώς ε, νόμους έχει κάθε χώρα. Εν πάση περιπτώσει μπορείτε να μας πείτε ίσως δύο λόγια γι' αυτό. Όσον αφορά το έτος ενεργούς γύρανσης, active aging, ε, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για την μακροχρόνια περίθαλψη ε, των ηλικιωμένων, την κακομεταχείριση, την κατάχρηση φαρμάκων κτλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη και μετά κυρία Μωρά. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ σήμερα. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή το φιλόδοξο πρόγραμμά σας και σκέφτηκα ότι ως εκπρόσωπος της Κομισιόν σήμερα εδώ ε, έχετε δύο χέρια. Ό,τι μας δίνετε με το ένα χέρι μας το παίρνετε με το άλλο μας δίνεται πάρα πολύ ωραία σχέδια, πάρα πολύ ωραία προγράμματα, αλλά όταν κοιτάζω την σύσταση για τη χώρα μου, την Ελλάδα, όταν φέρνω στο μυαλό μου την πραγματικότητα που επικρατεί ειδικά σήμερα, τη σημερινή μέρα, σκέφτομαι ότι βάζετε στόχους αλλά δεν μας βοηθάτε, δεν μας δίνετε τα εργαλεία για να μπορέσουμε να τους κατακτήσουμε. Όταν μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας, ένα παράδειγμα, αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Μία κυβέρνηση προσπαθεί και προσπαθεί κόντρα στην ιδεολογία της και έχει να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Εσείς εκεί, στο σημείο αυτό, βάζετε κι άλλη πίεση. Και τότε σκέφτομαι, οι αριθμοί που αναφέρατε, 23 εκατομμύρια άνεργοι, 113 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες στο κατόφλι της φτώχειας. Σε αυτούς πόσοι ακόμη Ευρωπαίοι πολίτες, Έλληνες πολίτες, Ισπανοί πολίτες, Πορτογάλοι πολίτες, Ιρλανδοί πολίτες θα προσθεθούν εάν η Κομισιόν συνεχίζει να πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι κυβερνήσεις κάνουν προσπάθειες και νομίζω ότι τις αξιολογείται αλλά πέρα από την, να, να τις αξιολογείτε χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μόρα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα το μεσημέρι μαζί μας. Είπατε ότι πρώτος μοχλός ε, πολιτικής σας είναι η καταπολέμηση της ανεργίας ε, και δι της ανεργίας των νέων. Είναι αληθές ότι σήμερα σχεδόν ένας στους πέντε νέους είναι και λέτε ότι θέλετε εσείς να βελτιώσετε την ποιότητα της εκπαίδευσης για να καταπολεμήσετε το, αυτά τα ποσοστά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι για τα άτομα που είναι τα πλέον ενδεοί και αυτούς που δεν επιτυγχάνουν είναι όχι ε, πιο ποιοτική εκπαίδευση αλλά ατομικευμένες, εξατομικευμένες απαντήσεις ε, στον τομέα της εκπαίδευσης για άτομα τα οποία ολοκληρώνουν τις σπουδέ τους χωρίς να έχουν κάποια ειδίκευση. Δεν ε, καταλαβαίνουν ολοκληρώσεις, δεν καταφέρνουν ολοκληρώσουν τις σπουδέ τους, αποτυγχάνουν. Δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω, είναι η διάρθρωση μεταξύ της εκπαίδευσης και της ε, εργασίας, η περίοδη άσκησης, μαθητείας. Καλή στόχη είναι, αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να δεσμευθούν και να ε, κάνουν μια δουλειά ανά επαγγελματικό κλάδο, διερευνητική δουλειά. Δηλαδή να δούμε το χρόνο της εκπαίδευσης ε, που είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον χώρο της άσκησης στην επιχείρηση. Θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή ώστε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση στα προγράμματα ανάπτυξης ε, των θέσεων διότι αν δεν γίνει αυτό θα εξακολουθήσουμε να χάσουμε τον τελικό μας στόχο. Τρίτο σημείο, πολύ γρήγορα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τα δύο αυτά εργαλεία πρέπει να διατηρηθούν. Το χρειαζόμαστε για να καταπολεμήσουμε ακριβώ την ανεργία και για να μπορέσουν οι πλέον ενδεεί και βρισκόμενοι σε μειονεκτική θέση να επανενταχθούν. Μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεν μιλήσατε όμως για το Ταμείο Προσάμβλησης στην Παγκοσμιοποίηση. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Τέλος να πω ότι μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ότι φαίνεται πολύ γρήγορα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις γιατί περιμένουν πολλοί οι πολίτες ε, και οι επιχειρήσεις ε, και οι εργαζόμενοι και βέβαια για τον τομέα της υγείας. Πολλά πρέπει να γίνουν πάνω σε αυτό το θέμα Πρέπει να τα κάνουμε και γρήγορα αλλά και με αποτελεσματικό τρόπο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, υπήρξαν συγκεκριμένα πολύ ακριβή ερωτήματα. Θα σας έλεγα λοιπόν να λάβετε τώρα το λόγο, αλλά έχουμε και μια συνάντηση με το Συμβούλιο και δεν μπορούμε να τους κάνουμε να περιμένουμε πολύ, άρα πρέπει να είστε κι εσείς λίγο σύντομος και ακολουθεί και άλλος γύρος ερωτήσεων. Σας παρακαλώ να είστε σύντομος, σαφής και ακριβής. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι σχετικά γρήγορος. Όμως είναι πράγματι πολύ μεγάλα τα προβλήματα. Θέλω να τονίσω μια πολύ σημαντική πτυχή της κρίσης πέραν του γεγονότος ότι έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις για τις κοινωνικές συνθήκες και την απασχόληση. Η Ευρώπη είναι πλέον περισσότερο διηρεμένη και υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες από ό,τι κατά το παρελθόν. πραγματικά υπάρχουν ε, φρικτά πράγματα που συμβαίνουν ε, ε, σε κάποιες χώρες. Υπάρχει μια γενική τέτοια κατάσταση και περιγραφή, αλλά αν γίνει κάτι καλό, παραδείγματο χάρη στη Γερμανία που έχουμε επίπεδα ρεκόρ απασχόληση στην Ολλανδία και στην Αυστρία που αντιμετωπίστηκε η κρίση με αρκετά χαμηλά ποσοστά ανεργίας, ούτε αυτό αναφέρεται. Φυσικά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα ή στην Ολλανδία είναι πρωτοσέλιδο αμέσως. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα, δηλαδή πιο πολύ τα αρνητικά πράγματα ε, προσελκύουν τους προβολείς της δημοσιότητας. Ε, πρόκειται για οξύτατη κρίση που βιώνουν ορισμένες χώρες και αυτός είναι ο λόγος ε, που συζητούνται και τα θέματα αυτά σε μεγαλύτερο βάθος. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει γενικευμένη πολιτική λιτότητας λόγω αυτών των θεμελιωδών αδυναμιών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, βλέπουμε τώρα να, αντιμετωπίζονται, να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες χώρες, συγκεκριμένες κρίσεις που απαιτούν συγκεκριμένη μεταχείριση, συγκεκριμένους χειρισμούς. Αλλά δεν έχουμε μία λύση που να είναι κοινή για όλες τις περιπτώσεις. Για την περίπτωση της Ισπανίας συγκεκριμένα να πω ότι σήμερα συνάντησα ε, τον Υπουργό Γκόμες και συζητήσαμε διάφορα θέματα. Η Ισπανία είναι μια σημαντική χώρα γιατί έχει την μεγαλύτερη ανεργία και τη μεγαλύτερη ανεργία ε, μεταξύ των νέων και βιώνει και αυτή μια περίοδο αστάθειας. Αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ευρεία ε, συνεννόηση και κατανόηση για το τι πρέπει να γίνει και το ίδιο ε, αφορά, ισχύει για την μεταρρύθμιση του κοινωνικού διαλόγου. Η κυβέρνηση της Ισπανίας πραγματικά είναι προσιλωμένη σε αυτό το στόχο και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα υποβάθμισης του κοινωνικού διάλογου από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, περί του αντιθέτου πρόκειται. Αυτό που θέλουμε είναι η ενίσχυση και παγίωση του κοινωνικού διαλόγου. Γιατί δεν είναι ένα μέσο κοινωνική σταθερότητα μόνο, αλλά είναι και ένα πλεονέκτημα για την οικονομία. Απλά πρέπει να υπάρξει ένα είδο ε, εξορθολογισμού, streamlining και πρέπει να βρεθεί ένας χώρος ε, ε, για, τις, ε, για τον κοινωνικό διάλογο στη διαπραγμάτευση των νέων συλλογικών συμφωνιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φτώχεια, τις κοινωνικές δαπάνες, εμβληματικές πρωτοβουλίες, συστάσεις, ειδικέ ε, κατά χώρα κτλ. Πρέπει να πω ότι οι χώρε φυσικά και δεν έχουν όλε το ίδιο φορολογικό περιθώριο ελιγμού. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώ. Γίνεται υποεκμετάλλευση του σε διάφορε χώρες, ε, ε, παραδείγματο χάρη στη Ρουμανία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την απορρόφηση των κονδύλιων ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όχι γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια ή γιατί είναι περιοριστική η Κομισιόν, αλλά λόγω έλλειψης ικανοτήτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων από τις εθνικές κυβερνήσεις σε σχέση με τις κοινωνικές δαπάνες. Παραδείγματο χάρη ε, υπάρχουν κάποια αιτήματα μεταφοράς κονδυλίων ε, στο πλαίσιο του ΕΚΤ ε, για σε ό,τι αφορά τα έργα οδοποιίας. Πάντως εγώ δεν συμφωνώ. Οι υπηρεσίε μου στην Ελλάδα, για παράδειγμα, εργάζονται πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να βρούμε μια καλύτερη χρήση των κονδυλίων του κοινωνικού ταμείου και να βοηθηθούν ειδικά ε, ομάδες που ήδη έχασαν ε, τη δουλειά τους ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του πολύ λιτού προπολογισμού ιδίως για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Σε ό,τι αφορά τώρα το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, και αυτό είναι σημαντικό ταμείο, ίσω μικρότερο σε μέγεθο μεν, αλλά εξίσου σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, όπω και το Κοινωνικό Ταμείο, ιδίω σε περιπτώσει έκτακτη ανάγκη ε, όταν έχουμε μεγάλη κλίμακα ε, απώλειες θέσεων εργασίας. Και πρέπει να σα πω ότι εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή διευθέτηση για το Ταμείο αυτό σε επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ. Να σα πω όμω ευθύ εξ δεν είναι εύκολο. Ε, το έχω πει και στο Κοινοβούλιο, έχω εκφράσει τις απόψεις μου, πρέπει ε, να πω ότι συνάδουν με τις γενικές γραμμές της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ταμείο αυτό. Ελπίζω λοιπόν και στην προσεχή περίοδο να είναι ακόμα πιο λειτουργικό επιχειρησιακό το Ταμείο αυτό και να λειτουργεί ταχύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Σε ό,τι αφορά την, ε, το θεματολόγιο της ασφάλειας στην εργασία, δεν θα ε, κάνουμε κάποια περαιτέρω πρόταση αν δεν δούμε ότι έχει ένα πρόσθετο, μια προσθέμενη αξία να προσφέρει. Υπάρχουν διατάξεις στην ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ε, μυοσκελετικέ διαταραχέ, ε, θέλουμε να υπάρχει συνέπεια. Θέλουμε να υπάρχει συνεκτικότητα με τα εφιστάμενα νομοθετικά μέσα που ισχύουν και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ενδεχομένω όμω να υπάρξουν και νέα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά το κάψμα, είναι σημαντικό αυτό και είναι γεγονός ότι έχει επιτευχθεί η πρόοδος στα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να σας δώσω τώρα το ακριβές νούμερο, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη ήδη έχουν κάποια μορφής, κάποια μορφής νομοθεσία για την κατάργηση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας, που ίσως να μην είναι ε, πλήρης απαγόρευση, να μην καλύπτεται το σύνολο των ε, χώρων εργασίας για την, ε, ε, τη βιομηχανία του catering και ώστε να υπάρχει κάποιες διαφορετικές διατάξεις. Όπως είπα, ίσως ε, ληφθεί σχετική πρωτοβουλία, θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα διαπιστώσουμε στην ε, προσεχή χρονική περίοδο. Ίσως όμως για του χρόνου θα είναι θα αιτιολογηθεί, το να περάσουμε σε αυτή την οδηγία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλού ομιλητέ. Θέλω να δώσω το λόγο σε όλους, γι' αυτό θα περιορίσω σε ένα λεπτό το χρόνο αγόρες στον καθένα. Η κυρία Σόετερ, η κυρία Σουέτερ, μετά κύριος Πουπάκης. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για την παρουσίαση του προγράμματος της Επιτροπής. Με ενδιαφέρει και πάλι για άλλη μια φορά αυτό το οποίο είπατε για τις θέσεις απασχόλησης. Είπατε ότι θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση. Τι βρίσκεται πίσω από αυτό. Θα είναι μια ανακοίνωση της Επιτροπής, θα είναι μια πράσινη βίβλος, ένα πρόγραμμα, πολιετές πρόγραμμα. Ενδιαφέρομαι να μάθω επακριβώς περί τίνος θα πρόκειται. Και το δεύτερο που είδα να απουσιάζει στα όσα μας είπατε είναι δηλαδή η απόσπαση εργαζομένων τι πρόκειται να γίνει. Εφέτος πρόκειται να υποβληθεί κάτι. Ο κύριος Μπαρόζο είχε πει ότι κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής θητείας θα υπεβάλλεται αυτό. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να προταθεί και πώς. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει ανάγκη η οδηγία αυτή να αλλάξει ώστε τα κενά που υπάρχουν και οι ελλείψεις σε σχέση με την απόφαση του 10, την ομολογία του 10 να καλυφθούν. Ποιες είναι οι προτάσεις σας σχετικά. Ο κύριος Πουπάκης και μετά η κυρία Γκιάρλινγκ. Είναι φανερό ότι η πρώτη προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας δεν έφερε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα με αποκλήσει των στόχων σε όλα σχεδόν τα μεγέθη. Έλλειμμα, έσοδα κρατικέ δαπάνε, καθυστερεί στην υλοποίηση των διαφορετικών αλλαγών, ανεργία να καλπάζει, απειλώντα τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και την ύφεση τη ελληνική οικονομία να βαθαίνει. Ξεκαθαρίζοντα σε κάθε περίπτωση ότι η λήψη μέτρων είναι αναγκαία σε κάθε περίπτωση για την αποκατάσταση τη σταθερότητα τη τα συγκεκριμένα όμω μέτρα που ελήφθησαν, στην ουσία πλήττουν κύρια τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε, εντείνουν τη φτώχεια και παράλληλα οδηγούν σε αδιέξοδο τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή με έντονε αντιδράσει που βλέπουμε καθημερινά των πολιτών, όπω εκδηλώνονται με τι πρόσφατε μαζικέ κινητοποίησει σε όλη τη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν απλά την εκτίμησή σα. Μήπω θα ήταν σκόπιμη στο πλαίσιο των συστάσεων η αναθεώρηση κάποιων σημείων του μνημονίου στην κατεύθυνση διασφάλιση επιτυχία στου δημοσιονομικού στόχου στη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξη για νέε θέσει απασχόληση, αναγκαία αποκατάσταση των κοινωνικών ανισορροπιών και ενίσχυση τη αξιοπιστία στη χώρα στι διεθνεί χρηματαγορέ. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη ε, διαρκεί πλέον τρία χρόνια. και περνάει σε όλες τις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το αναφέρατε ακροθυγώς, αλλά δεν είδαμε αν κάπου έχουμε και επιτυχίες. Έχουμε μεγάλα ποσοστά ανεργίας, κυρίως δε στους νέους και αυτά τα ποσοστά είναι μεγάλα σε όλες τις χώρες. Νομίζω όμως ότι ε, θα πρέπει να αναλύσουμε κάπως ε, το τι ε, μέτρα έχουν πάρει οι χώρες μέλη, αν λειτουργούν τα μέτρα αυτά. Εγώ θα πω δύο λόγια για το Ηνωμένο Βασίλειο, που οπωσδήποτε ε, αντιμετωπίζει ε, σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα και, μεγάλες, και μεγάλα οικονομικά διακυβεύματα. Ε, υψηλό ποσοστό ανεργίας, το υψηλότερο για, και με μεγάλη αυξητική τάση μάλιστα επί πολλούς μήνες, το υψηλότερο ποσοστό τα πολλά, για πολλές δεκαετίες. Επομένως, που έγκυται η διαφορά, η ευελιξία ε, της ε, ευελιξία της ε, αγοράς ε, εργασίας. Δηλαδή ε, είχαμε προβλήματα και τη δεκαετία του 80, αλλά όμως τα πράγματα τότε αντιμετωπίστηκαν με πολύ καλύτερο τρόπο, γιατί πλέον τη μεταρρυθμίσαμε την αγορά και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά τέτοιες κρίσεις. Ο χρόνος εργασίας, ένα σημαντικό θέμα, πολύ σημαντικό. Δυστυχώς μιλάει και η Πρόεδρος μαζί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Το, ρόλο έχει, το λόγο έχει ο Αυτά που είπατε για το πρόγραμμα εργασίας όμως ε, για την κοινωνική εταιρική ευθύνη θα πρέπει να δούμε και αυτή η σημασία της παράλληλα με τις άλλες πρωτοβουλίες σας σε σχέση με θέματα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε παραδείγματα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τα δάνεια και τις πιστώσεις σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δούμε εδώ και σε σχέση με τα δίκτυα τα οποία υπάρχουν στην Βρετανία πώς αξιολογείται την εξέλιξη εκεί και σε χώρες πέρα από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι πρόβλημα το να υπάρχουν ξεχωριστά προγράμματα σε σχέση με τους νέους αν δεν υπάρχουν ευκαιρίες ε, ως θέσεις απασχόλησης για να απασχοληθούν. Ποια νομίζετε ότι είναι η καλύτερη αντίδραση και πρωτοβουλία σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Ράκκιν παρακαλώ και μετά Μπάουερ. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι έχετε ένα φιλόδοξο σχέδιο και όπως ε, είπατε πρέπει να έχουμε αξιόπιστες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να προσφέρουμε λύσεις. Και εκείνο σε σχέση με τις προκλήσεις ε, και αναφέρατε πρόκληση 23 εκατομμύρια ανέργους και χρησιμοποίησατε τον όρο freaky horror που είναι επακριβής για αυτή την κατάσταση που μας ξεπερνά όλους. Πολύ ανησυχώ για τους ε, ανέργους και είπατε ότι κάποιες χώρες έχουν ε, προ, ε, προϋπολογισμούς δημοσιονομικής λιτότητας, άλλες όχι. Έχουμε όμως απώλειες θέσεων απασχόλησης και στις υπηρεσίες και πρέπει εδώ να δούμε ε, την προώθηση πολιτικών για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Είπατε για τα καλά μαντάτα από τη Γερμανία και την Αυστρία. Δεν είπατε όμω ότι έχουν μεγάλα πλεονάσματα αυτέ τι χώρε. Άλλε χώρε έχουν μεγάλα μ, ε, ελλείμματα και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα. Μου φαίνεται ότι βλέπει τα ελλείμματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν βλέπει τα πλεονάσματα σε σχέση με την αντιμετώπιση των προβλημάτων μα. Και έτσι λοιπόν με χαρά βλέπουμε το πρόγραμμα εργασίας. Όμως πιστεύω ότι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μπάουερ, μετά ο κύριος Κοφεράτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι τον τελευταίο καιρό είδαμε ότι υπήρξε τροχοπέδηση στο Συμβούλιο σε σχέση με την οδηγία για τις ε, άδειες, ε, γονεϊκές άδειες ε, για άνδρες, πατέρες και γυναίκες. Τι προτείνει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναδιατυπώσει αυτή την πρόταση ή θα υποβάλει μια νέα πρόταση οδηγίας. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας εκπλήσει Υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια που ζουν στη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι μειώνεται, θα μειωθεί ο αριθμός των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, θα εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για μια ανάπτυξη που ενσωματώνει και εντάσσει αυτούς του ανθρώπους. Ο κύριος Κοφέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με πολύ μεγάλη υπομονή άκουσα τις, ε, ε, και διάβασα τις ε, ενδείξεις και συστάσεις ε, προς ε, τα κράτη-μέλη από πλευρά της Επιτροπής σας βεβαιώ ότι δεν κατάφερα να βρω κοινό πεδίο γιατί άλλα λέει στη μία χώρα άλλα λέει στην άλλη ας πούμε για την χώρα μου λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έτσι μια διτότητα του και μια διαδικότητα στην αγορά ε, εργασίας, ε, κάνει μια πρόταση η οποία δεν είναι καθόλου λογική ε, και στις συστάσεις της Επιτροπής υπάρχει και μία σύσταση για το πώς θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συλλογικές συμβάσεις και οι προτάσεις που κάνετε για αυτή την τροποποίηση ε, των συλλογικών συμβάσεων μπορεί να εφαρμοστεί μονάχα σε ελάχιστες ε, ε, επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Γκουτιέρες και μετά η κυρία Εγκικούξη. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένας όρος που είναι του σειρμού στις μέρες μας. Η μεταρρυθμιστική κόποση τη γέννησαν αυτή την έννοια οι αγορές σε σχέση με τους στόκους ε, και με, την, ε, με το χρέος. Κατά την άποψή μου, στις συστάσεις που έχει εκπονήσει η Κομισιόν προς τα διάφορα κράτη-μέλη, που έχουν υποτίθεται ότι έχουν ε, μία κόποση σε σχέση με την έμπνευση για την εξέβριση λύσεων, ταυτόχρονα λέγεται ότι σε ό,τι αφορά την ε, λιτότητα ή σε ό,τι αφορά την οικονομική εξυγένση. Ουσιαστικά οι ίδιες συνταγές δίνονται, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόταση για την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Λέει η Κομισιόν ότι θα πρέπει να ε, γίνει μεγαλύτερη εργασιακή μεταρρύθμιση για να ενισχυθεί η αγορά εργασίας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Ε, ρυθμίζεται η αγορά μεν, αλλά ανάπτυξη δημιουργείται μόνο με την ε, δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να πω συγκεκριμένα με τη χώρα μου και τι κοινωνικέ ε, εισφορέ βλέπουμε ότι το δίκτυο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες καταραίει, διότι τα μέτρα είναι ε, ανυπόστατα. Λένε ότι θα βελτιώσουν τις κοινωνικές ε, συνθήκες και τις κοινωνικές περιτάσεις, αλλά τελικά μας λένε ότι πρέπει να μειώσουμε τις συντάξεις, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν υπάρχουν ε, αρκετοί πόροι να στηρίξουν τα ταμεία. Θα ήθελα τρία λεπτά για να πω έστω κάτι που να έχει νόημα. Ε, πρόεδρος, ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη και από τους βουλευτές και από τον Επίτροπο γιατί ε, δυστυχώς πήρε μεγαλύτερο χρόνο η πρωινή μας συνεδρία και πραγματικά είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο και απογοητευτικό το όλο εγχείρημα και εγώ που ήθελα να κάνω ερωτήσεις για την εξόριση κατάσταση της δικής μου χώρας αλλά και άλλων χωρών και δεν θα τις κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Κυρία Κίνγκα Γκέντς είναι τελευταία ομιλήτρια. Ναι, κατάλαβα ότι είναι πολύ μικρός ο χρόνος για τη συζήτηση και εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα διπλά μηνύματα στρατηγική για τους Ρωμά, πρόγραμμα στο πρόγραμμα εργασίας και από την άλλη πλευρά συγκεκριμένες συστάσεις ε, κατά χώρα που δίνουν την εντύπωση ότι σε κάποια χρόνια η Ευρώπη θα είναι πολύ διαφορετική από την Ευρώπη των τελευταίων ετών. Πολύ λιγότερη κοινωνική Ευρώπη θα είναι. Το ερώτημά θα ήταν, ξέρω ότι δεν είναι πολύ ο Πώς βλέπετε αυτή τη μελλοντική Ευρώπη με βάση τις συστάσεις αυτές ε, κατά χώρα, πώς τα βλέπετε αυτά τα δύο να συνάδουν, να συμφιλιώνονται το ένα με το άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πρέπει να συναντώμαστε όσο σε πιο τακτικά διαστήματα να καλλιεργούμε τις συζητήσεις και επαφές μεταξύ μας και όσο το δυνατόν να καλλιεργούμε αυτές τις συζητήσεις σε μεγαλύτερο ή στενότερο κύκλο. Σε σχέση με τις πρωτοβουλίες για την Ευρώπη θα ήθελα να αποφύγουμε του να μιλάμε, το να μιλάμε για την κρίση στην ε, Ευρώπη και να βλέπουμε την Ευρώπη σαν μια ιδανική περίπτωση. Πριν από την κρίση είχαμε μια περίοδο ευημερίας χωρίς όμως την άρση, την εκρίζωση της ε, φτώχειας. Ε, κάποιες χώρες είχαν θετικές πολιτικές ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο Ρίτσαρντ αποτελεσματικές πολιτικές για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και για την ένταξη των φτωχών και ελπίζω ότι οι δημοσιονομικές περικοπές δεν θα πλήξουν τέτοιου είδους πολιτικές ή τα αποτελέσματα που είναι θετικά. Όμως η κρίση μεταμορφώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι όχι μόνο η κρίση, αλλά και εμείς οι ίδιοι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και να μεταρρυθμίσουμε και να μεταμορφώσουμε την κοινωνία και την οικονομία μας και να κάνουμε την κοινωνία και την οικονομία πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουμε τη συνεκτικότητα και συνοχή και την ε, κοινωνική διάσταση, να την ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο. Αν μειώσουμε μόνο τον αριθμό κατά 20 εκατομμύρια των φτωχών ήδη θα έχουμε πετύχει κάτι ως ένα πρώτο βήμα. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το στόχο ήταν ήδη και πολύ δύσκολο. Πέρυσι για παράδειγμα να μετρήσουμε και να σταθμίσουμε τι είναι φιλόδοξο και ρεαλιστικό ταυτόχρονα στο ευρωπαϊκό επίπεδο με εμπλοκή όλων των κρατών μελών δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Το κλειδί είναι να διασφαλίσουμε ότι θα, θα αντιστρέψουμε την τάση. Βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με την ε, μεγαλύτερη ε, ανισότητα και την πρόσφατη ε, περίοδο υπήρξε σε σχέση με την, ε, εκείνους που βρίσκονται στο κατόφλι της φτώχειας και ζουν σε αποκλεισμό υπήρχε ένα είδος άγνοιας. Πρέπει να μπορούν να μετρηθούν τα αποτελέσματα, όχι μόνο σε σχέση με το 2020 που είναι η καταληκτική ημερομηνία, αλλά και με μια ενδιάμεση αναθεώρηση για να δούμε αν θα υπάρξει μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε ήδη τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη για την φτώχεια και την απασχόληση και δεν καταλήγουν σε αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει πανευρωπαϊκά στην Ευρώπη πέρυσι. Αυτά που μπορώ να πω λοιπόν είναι, αν διατηρήσουμε τους φιλόδοξους στόχους και εργαστούμε για να υπάρξει μια δυνατότητα αναθεώρησης και αναβάθμισης ε, στο μεσοδιάστημα σε μια ενδιάμεση αναθεώρηση, καλό θα είναι αυτό. Δύο λόγια για το νομοθετικό έργο, γιατί τέθηκε μια ερώτηση για το χρόνο απασχόλησης και την απόσπαση εργαζομένων. Δεν ανέφερα το θέμα αυτό για την απόσπαση posting και θα το κάνουμε φέτος. Και όπως είχαμε προαναγγείλει στην ε, πράξη για την ενιαία αγορά, από τον Επίτροπο Μπάρνιε, θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία αυτή και είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι κατά τα τέλη αυτού του μήνα θα υπάρξει μια διάσκεψη με τον ήδη τη συμμετοχή του κυρίου Μπαρνιέ και εμού και θα υπάρξει και συμμετοχή άλλων όπως ε, και της κυρίας Προέδρου και μετά από αυτή τη διάσκεψη τη σύνοδο αυτή θα αναλυθεί μια νέα πρωτοβουλία και θα υπάρξει μια νέα οδηγία όσον αφορά τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα που θα ενταχθούν ε, και θα παρουσιαστούν όσον αφορά ε, την ιστερότερη φάση του έτους αλλά και για την απόσπαση εργαζομένων. Όπως θα γνωρίζετε βρισκόμαστε, ε, εμπλεκόμαστε υπέρ των κοινωνικών εταίρων στο ευρωπαϊκό επίπεδο εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των ε, εργοδοτών είπαν ότι είναι πρόθυμοι να διαβουλευτούν. Συζητούν για ένα πλαίσιο και για το εύρος ε, προτού υπάρξει η επιβεβαίωση και υπάρξει η πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτές τις διαβουλεύσεις και τις επιτροπής. Γίνονται διαπραγματεύσεις για το χρόνο, την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Χαίρομαι για το ότι το κάνουν αυτό και με χαρά βλέπω ότι και οι δύο έχουν επικοδομητικό πνεύμα να καταλήξουν σε θετικά συμπεράσματα και μέχρι ότου απευθυνθεί αυτή η πρόσκληση να εμπλακούμε και εμείς δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια για αυτό το θέμα. Για τις πράσινες ε, θέσεις απασχόλησης προετοιμάζουμε ένα πράσινο βιβλίο που είναι η πιο εύθετη, ο πιο σκόπιμος τρόπος να καλύψουμε αυτό το θέμα. Είναι και μια καλή ευκαιρία για να προσκαλέσουμε να υποβληθούν προτάσεις και σχόλια γιατί βρισκόμαστε ευθυγραμμισμένοι με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και με άλλους ε, ορισμούς, αλλά θέλουμε να έχουμε επαρκείς προτάσεις από πλευράς της Ευρώπης που θα μπορούν να ενταχθούν και ιδέες. Αυτό είναι καλό, αφενός για να βοηθήσουμε να ε, εξειδικεύσουμε σε λεπτότερο βαθμό τις πολιτικές μας για την απασχόληση αλλά και για την εμπλοκή και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με πολλά από τα προγράμματα που θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μετάβαση όσον αφορά μια πιο αποτελεσματική οικονομία για την Ελλάδα. Δύο λόγια. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτά που έκανε η κυβέρνηση διότι κληρονόμησε ως κληροδότημα μια πραγματικά απίστευτη οικονομικά, δύσκολη στην αντιμετώπιση της οικονομική κατάσταση. Σκληρά μέτρα έπρεπε να ληφθούν που ήταν κατά της ίδιας της δημοφιλίας της κυβέρνησης, αλλά έκαναν ό,τι ήταν το καλύτερο υπέρ της Ελλάδας και παραμένουν ένα σεβαστό μέλος της ε, ε, Ευρώπης ε, και της ζώνης ευρώ. Όμως αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία αυτόματου πιλότου, αυτόματης πορείας. Ιδιαίτερα όταν συντάχθηκε το ελληνικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της Ελλάδας δεν υπήρχε τότε η Ιρλανδική κρίση ούτε η κρίση της Πορτογαλίας. Έχουν αλλάξει τώρα οι συνιστώσεις εκβάθρων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο συνάδελφός μου όλοι Ρένο Επίτροπος αλλά και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδιαίτερα και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου όλοι να εξετάσουν με ένα νέο βλέμμα, με μια νέα καινούρια ματιά αυτή την νέα κατάσταση και να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής της ε, Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ε, και την βοήθεια της Ελλάδας. Ίσως αυτό το οποίο λείπει, απουσιάζει, είναι μια στρατηγική για την ανάκαμψη και την αναδόμηση, αναδιάθρωση της ευρωπαϊκής οικονομίας που θα αποκαθιστούσε την εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό φυσικά απαιτεί μια ισχυρή και αξιόπιστη πολιτική διαχείριση, διακυβέρνηση και πιστεύω ότι μπορεί, είναι σε θέση η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει να τα ε, πηγαίνει καλά, να έχει καλές επιδόσεις. Από κοινού με, το, με άλλους επιτρόπους και τον Αντιπρόεδρο κύριο Ταγιάννη και τον κύριο Μισελ Μπανιέ, από κοινού πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν προτάσεις που θα ε, διατυπωθούν όσον αφορά την πλευρά της απασχόλησης για την CSR στο Όσλο να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι μόνο ένα, μια ευρωπαϊκή προσπάθεια αλλά που θα έχει και μια πολύ ισχυρή ε, παγκόσμια οικουμενική συνιστόσα όσον αφορά και τις επιχειρήσεις ε, που βρίσκονται εκτός Ευρώπης ε, οικουμενικά. Δεν θα είναι μόνο το θέμα της Ευρώπης ε, που πρέπει να δούμε και να επικεντρωθούμε σε αυτό αλλά και παγκόσμια να δούμε πώς θα υπάρξει η σωστή τοποθέτηση και δράση αλλά αυτό θα πρέπει να ε, το δουν οι υπεύθυνοι σε σχέση και με την κοινωνική διάσταση για την παγκοσμιοποίηση και σε σχέση με την ε, ατζέντα της ε, CSR πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη μαζί με την κοινωνική διάσταση και την παγκοσμιοποίηση. Προφανώς δεν μπορώ, δεν μπορώ πολλά άλλα θέματα να καλύψω και να επεκταθώ επί παντός του επιστητού κάναμε βήματα προς τα εμπρός, σημειώθηκε πρόοδος πιστεύω. Ήδη τα πρώτα βήματα υπάρχουν, είναι δεδομένο και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Υπάρχει βέβαια ανάγκη να επανορθωθούν, να αντισταθμιστούν οι διαρθρωτικές μη ισόρροπες σχέσεις και δυσαναλογίες προτού μπορεί να διασφαλιστεί ότι στον επόμενο κύκλο θα υπάρξει ισχυρότερη έμφαση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, πράγμα το οποίο είναι ευκταίο και χρειάζεται ιδιαίτερα πρέπει να ξεκινήσουμε έγκαιρα αυτή την ε, εκστρατεία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα αντανακλώνται περισσότερο οι ανάγκες ε, της ε, σωστής ανάπτυξης, μια σωστής ισορροπίας για την επίτευξη της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις μαραθώνιες παρεμβάσεις αλλά δυστυχώς πρέπει να ε, σταματήσω η συνεδρίασή μας. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους που τους πίεσα και αυτούς που δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο ή να έχουν όλο το χρόνο που ήθελαν για τις ερωτήσεις τους. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Θα τα ξαναπούμε στην προσεχή συνεδρίαση συγκεκριμένα στις 11 Ιουλίου, λέει η Πρόεδρος. 11 Ιουλίου.